θα γίνει στο τέλος των συζητήσεων. Ακολουθεί το θέμα του Νεπάλ. Θα ζητήσω πρώτα απ' όλα από τους ε, συντάκτες να λάβουν τον λόγο και πρώτα απ' όλα η κυρία Γκέριγκερντε Εντενμπεργκ. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει για το Αμερικανικό Σύνταγμα πως το Σύνταγμα δεν εγγυάται την ευτυχία μόνο την επιδίωξή της. Σήμερα λοιπόν οι Νεπαλέζοι δεν έχουν ούτε αυτή την δυνατότητα. Συνεχίζεται η σύνταξη του συντάγματος και οι μαοιστές και οι κομμουνιστές δεν είναι διατεθειμένοι να συμβαστούν. Το δε ο δε στρατός είναι μυστικοπαθής. Από την άλλη πλευρά του φάσματος 30 ε, εκατομμύρια πολίτες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ζουν σε φτώχεια, χωρίς ηλεκτρισμό και βεβαίως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα ισχυρά του σημεία που είναι η γεωγραφική του θέση. Τον ΕΠΑΛ ζητάμε λοιπόν και την τήρηση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του 2008 και την ψήφιση ενός νέου συντάγματος που θα προστατεύει τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα αντιπροσωπεύει κάποια πρόοδο για τη δημοκρατία στο Νεπάλ. Ω ευρωβουλευτή μια χώρα που είχε διχαστεί πολλέ φορέ στο παρελθόν, αντιλαμβάνομαι το τι περνάει το Νεπάλ. Το Σύνταγμα δεν θα προσφέρει ευτυχία, αλλά θα του επιτρέψει να την επιδιώξουν. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, ο κύριος Τάνο ένα λεπτό. Η πολιτική αστάθεια του Νεπάλ δεν μας εκπλήσει. δεδομένου των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα. Ε, η εξέγερση του 2001 υπέσκεψε την μοναρχία και το κράτος απέτυχε στην καταπολέμηση του μαγιστικού κινήματος. Ε, πριν από δύο χρόνια έγινε αλλαγή στην κυβέρνηση και ε, από ό,τι φαίνεται η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ε, δεν έχει πετύχει. Ο λαός εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση φτώχειας και καταπίεσης. Ε, δυστυχώς ε, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη συμφιλίωση και ε, τη βελτίωση του, συστήματος, του δικαστικού συστήματος. Ελπίζω θα εστιαστούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα, δίνοντας και ανθρωπιστική βοήθεια. το Νεπάλ κινδυνεύει να αποτύχει ως κράτος συνολικά και να καταρρεύσει και θα δημιουργήσει σημαντικότητες πρόσθετες απλές για την ασφάλεια της Ασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Για δύο λεπτά ε, Ευχαριστώ. Ε, εκπροσωπώ τον Τζιν Λάμπροκ, ε, που είναι επικεφαλή τη αντιπροσωπεία ε, με αυτή τη χώρα δεν μπόρεσε να είναι παρούσα εδώ. Θα ήθελα να σα πω, να σα πει εκείνη μάλλον το εξή. Τα τελευταία χρόνια το Νεπάλ έχει κάνει θετικέ αλλαγέ, ε, όπως λέει και το ψήφισμα, ε, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ε, η κατάσταση όπως εξελίσσεται, εξελίσσεται ε, δημιουργεί προβλήματα για την εφαρμογή της Συνευτικής Συμφωνίας και ακόμη δεν έχει συνταχθεί το νέο σύνταγμα. Ε, επομένως δεν έχουν, προσπισ... δεν έχουν προωθηθεί τα... οι αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει τώρα η συντακτική συνέλευση. Προσπαθούν να κάνουν μια απόπειρα της τελευταίας στιγμής, ούτως ώστε να προωθήσουν την ειρηνευτική συμφωνία και την, το νέο σύνταγμα. Αυτό το εκλεγμένο σώμα έχει μία ευκαιρία να τα καταφέρει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, για πολιτική σταθερότητα. Υπάρχουν δυνατότητες για ε, εξέλιξη των νεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα είναι δύσκολες οι επενδύσεις χωρίς σταθερότητα. Η δημοκρατία και ε, το κράτος δικαίου πρέπει να εγκαθιδρυθούν στη χώρα αυτή η ένταξη των πρώην μαοιστών μαχητών ε, πρέπει να γίνει ε, και θα είναι και δείγμα ε, δημοκρατικής πρόοδου της χώρας αυτής. Θεωρούμε ότι η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουν με πρακτικό τρόπο αν χρειαστεί να βοηθήσουν τη χώρα αυτή. Θα είναι κρίμα όμως να αποσυρθούν οι δυνάμεις του ΟΗΕ αν δεν σημειωθεί πρόοδος τις επόμενες Νομίζω ότι πρέπει ε, το τριμερέ σχέδιο να προωθηθεί από όλου του ενδιαφερόμενου, αλλιώ θα υπάρξει εμπιστοσύνη του λαού. Ε, Όλε οι εξελίξει συνδέονται με την δυνατότητα πολιτική πρόοδου. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Φρεντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι ανισχυτική. Η βία αυξάνεται σε αυτή τη χώρα. Για να ενισχυθεί λοιπόν η διαδικασία συμφιλίωσης μετά τον εμφύλιο των 10 ετών που τελείωσε μόλις το 2006 και σκότωσε 13.000 άτομα χρειάζεται ένα νέο σύνταγμα. Έτσι θα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για την πολιτική ζωή στον Νεπάλ. Αν προωθήσουμε βεβαίως τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό θεωρώ πως τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διαπραγματευτούν χωρίς προϋποθέσεις για μια συντακτική συνέλευση. Όπως έχει δείξει η έκθεση του ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί και η δικαιοσύνη για να βρεθεί μια ειρηνική λύση στην σύγκρουση. Τέλος, να αναφέρω πως η πολιτική αστάθεια έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση του Νεπάλ που είναι μία από τις οχότερες χώρες. Ξέρετε, χωρίς σταθερότητα δεν υπάρχει ευημερία. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ο κύριος Χίγκινς για δύο λεπτά. Thank you, Chair. The Η φεοδαλιστική μοναρχία έπεσε το 2006 και αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα πρόοδου για το λαό. Η εργατική τάξη, η μέσια τάξη και οι αγρότες πέτυχαν αυτή τη νίκη με μαζικές κινητοποίησεις ε, του λαϊκού κινήματος. Είναι σαφές όμως πλέον ότι ε, η καπιταλιστική καθεστική τάξη ε, δεν επιθυμεί αυτή η επανάσταση να πάει πιο μακριά γιατί αυτό θα απειλούσε τον οικονομικό έλεγχο που έχουν και την προνομή θέση που κατέχουν στην κοινωνία. 50% των 29 εκατομμυρίων κατοίκων του Νεπάλ ε, ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 16% ε, από αυτούς ε, δεν διατρέφονται σωστά. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς γη και το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, έκανε το λάθος να εισέλθει στη, μετά το 2006 μαζί με κόμματα της δεξιάς σε κυβέρνηση, συμμαχική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνασπισμού ε, ε, κάτι που οδήγησε ε, στην, στην διατήρηση του ίδιου συστήματος με τη συνέχιση του καπιταλιστικού συστήματος. Ε, η γενική απεργία φέτος μετά τα γεγονότα του 2006 δείχνουν ότι η, ε, η εργατική τάξη και οι φτωχοί εξακολουθούν να ζητούν, να αναζητούν ένα μέλλον καλύτερο και χωρίς καταπίεση. Θα πρέπει τα κόμματα τα οποία πραγματικά αντιπροσωπεύουν τις μάζες να καταφέρουν να τεθούν επικεφαλής του αγώνα εναντίον του συστήματος και να προκειμένου να δημοσιοποιηθεί ε, ο, ο πλούτος που βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια και να εκδημοκρατιστεί το σύστημα, κάτι που θα οδηγούσε σε κοινωνικέ μεταρρυθμίσεις υπέρ των δεκάδων εκατομμυρίων φτωχών, όχι μόνο στην Επάλα αλλά και στην Ινδία και στην Κίνα. Ε, χρειάζεται επίσης να γίνει σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των διαφορών κοινοτήτων του Νεπάλ. Ευχαριστώ κύριε η κυρία Σάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Μετά από δεκαετίες ε, ε, φιλίου πολέμου ε, υπάρχει συμφωνία το 2006 μεταξύ των διαφόρων μερών, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει σταθερότητα. Χρειάζεται ένα σύνταγμα για τη δημοκρατία όμως επειδή υπάρχει αδιέξοδο στη συνταγματική συνέλευση, χρειάστηκε να παραταθεί η θητεία του για ένα χρόνο. Το Νεπάλ έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό για να αναπτυχθεί οικονομικά και να περιορίσει τη φτώχεια. Αλλά χρειάζεται σταθερότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχά, θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για την καταπάτηση των νόμων. Αυτό πρέπει να συμβεί. Ε, και τα μέλη του PLA και των ε, δυνάμεων ασφαλεία. Και ο ΙΕ θα πρέπει να παίξει το ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ε, σε διεθνεί ένοπλε δυνάμει. Θα πρέπει να υπάρξει να λάμψει αλήθεια, να υπάρξει συμφιλίωση για να αποδοθούν ευθύνε για όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Τα μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσουν το ώστε να υπάρξει ε, μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επίσης να εγκρίνουν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα θέλαμε ε, τα κρατη να υποστηρίξουν την ε, νεπαλέζικη κυβέρνηση και όλων των μερών, ούτως ώστε να αποκαταστήσουν και να ενσωματώσουν ε, τους μοριστές μαχητές ε, και να τους εντάξουν στο στρατό και να βρεθούν λύσεις για αυτούς που δεν μπορούν να ενταχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να απαγορεύσει την εξαγωγή ε, θανατηφόρων όπλων στο Νεπάλ καθώς και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση όπως ε, λέει το ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο σήμερα. Ευχαριστώ. Ήσασταν η τελευταία των συντακτών. Θα ακολουθήσουν οι ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ο έμφυλιος ε, πόλεμος ε, τελείωσε βέβαια το 2006 μετά από 10 χρόνια, αλλά η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη στο Νεπάλ. Χωρίς σταθερότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί το Νεπάλ, όπως οι γειτονές του, η Ινδία και η Κίνα μια συμμαχία 22 αντιμαοικών κομμάτων δεν μπόρεσε να υιοθετήσει το Σύνταγμα μέχρι το Μάιο του 2010, οπότε καλό είναι να παραταθεί κατά ένα έτος η εντολή της συντακτικής συνέλευσης. Είναι σημαντικό να υιοθετηθεί Σύνταγμα για να λειτουργήσει το κράτος δικαίου και να τηρηθούν τα δικαιώματα των πολιτών. Να τονίσω πως οι σημαντικότερες απειλές στη σταθερότητα του Νεπάλ είναι οι ακραίες απόψεις και η βία ως μέσο λύση των πολιτικών προβλημάτων. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου, ο κύριος Τζόμπρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στο Νεπάλ είναι ενσχετική εδώ και πολλά χρόνια πρώτες εκλογές έλαβαν χώρα το 1958. Παρ' όλα αυτά, το δημοκρατικό σύστημα δεν διέρχεσε για πολύ καιρό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούσαμε, παρατηρούσαμε κάποια πρόοδο. Το 2006 ε, μια συμφωνία, ειρηνευτική συμφωνία τέλειωσε, ε, έδωσε τέλος σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Κατόπιν έγιναν εκλογές ε, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πλην όμως τελευταία βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Και από ό,τι ε, φαίνεται, ε, η τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξουν τις ε, προσπάθειες ε, εδραίωσης τη ειρήνη και της σταθερότητα στη χώρα με τη διεύθυνση των αρμοδιοτήτων της συντακτική ε, συνέλευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσιόμπρο. Να παρακαλέσω όσους διαβάζουν κείμενα από μέσα να τα διαβάζουν κάπως πιο αργά γιατί δεν περνάει μετά και το περιεχόμενο. Ακολουθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θα διαβάσω. Θα μιλήσω ελεύθερα και μάλιστα αργά-αργά, παρότι αυτό αντιβαίνει στη φύση μου. Ε, παραδόξως η κατάσταση στο Νεπάλ βελτιώνεται. Χάρη σε, ποιε, σε κάποιες αποφάσεις να δοθεί περισσότερη εξουσία στο κοινοβούλιο. Το Νεπάλ όμως μόλις έχει ξεκινήσει ένα μακρό ταξίδι. Ο εμφύλιος πόλεμος έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη χώρα και μόλις τώρα αρχίζουν να βλέπουν οι άνθρωποι του Νεπάλ ε, το φως στο βάθος του τούνελ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά για να υποστηρίξει τη χώρα στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα αυτή έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα και τα οράματά τους και οι προτάσεις τους για μεταρρυθμίσεις ε, είναι κομμουνιστικές και μαοιστικές ε, και μάλιστα μερικές φορές αντιφατικές μεταξύ τους. Περνάμε λοιπόν στη διαδικασία και τη Κυρία Κόρολα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εμφύλιος αυτός πόλεμος ε, που κράτησε σχεδόν 10 ε, χρόνια στο Νεπάλ τελείωσε επιτέλους με μια ειρηνευτική συμφωνία. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση δεν είναι ήρεμη. Ο στρατός και τα πολιτικά κόμματα δεν ε, ελέγχουν την κατάσταση. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στο Νεπάλ, αναταραχές. Ε, το πρόβλημα αφορά την ηγεσία του στρατού και τον δημοκρατικό έλεγχο του στρατού. Ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καλή του δουλειά για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα και να έχει ασφαλές μέλλον τον ΕΠΑΛ. Ευχαριστώ η κυρία Κρετού. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ό,τι αφορά την ένταση και τη βία που επικρατεί στο Νεπάλ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα πιο οδυνηρά προβλήματα των Νεπαλέζων, τη φτώχεια. Ε, οι συνθήκες ε, ζωής είναι εξαιρετικά επισφαλείς και αυτό επιδεινώνεται από την πολιτική αστάθεια. Ε, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Η χώρα βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα σε δύο από τις πιο σημαντικές αναδυόμενες χώρες, την Κίνα και την Ινδία. Αλλά εξαιτία της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα δεν επωφελείται από αυτό σε οικονομικούς όρους. Το 1 τρίτο των κατοίκων του ε, ε, ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ο αλφαβητισμός είναι πάρα πολύ ψηλός υπάρχει σημαντική ενεργειακή έλλειψη ενέργειας, έλλειψη τροφίμων. Ε, η φτώχεια δημιουργεί και ανθρωπιστικά προβλήματα, όχι μόνο πολιτικές εντάσεις. Θα πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν στην ανάπτυξη και της οικονομίας του Νεπάλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρετού. Ο κύριος κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι τυχερός γιατί επισκέφθηκα πρόσφατα τον Νεπάλ. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε είναι πως η πολιτική διαδικασία στο Νεπάλ είναι εύθραυστη αλλά προχωρά. Είναι όμως παράλογο να συνεχίσει αυτή η διαδικασία χωρίς αφοπλισμό των μαοϊκών γιατί οι Μαοικοί δεν λαμβάνουν μέρος στην διαδικασία αυτή και θέλουν να αλλάξει κυβέρνηση χωρίς να αφοπλιστούν. Δεν γίνεται να υπάρχει πολιτική διαδικασία με κάποιους ενόπλους που δεν αφοπλίζονται και δεν είναι τα όπλα τους στις αρχές. Και μέχρι να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο πρέπει να πείσουμε ήπια και τις δύο πλευρές των ΕΠΑΛ πως είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον του, ναού, του λαού του Νεπάλ να αφοπλιστούν και να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ενότητας. Ευχαριστώ κύριε Ντίβα. Τελευταίος η κυρία Φοντούρν Χόενστάιν. Ε, για αρκετά χρονιά έχω, έζησα στο Νεπάλ. Την εποχή που οι Νεπαλέζοι πήραν την τύχη στα χέρια τους και προσπάθησαν να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα πριν από 20 περίπου χρόνια. Τότε ήμουν αισιόδοξη. Από ό,τι φαίνεται αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι κανείς θα φανταζόταν εκείνη την εποχή. Το Νεπάλ ε, είναι, έχει μια κουλτούρα πολύ παλιά, πολύ πλούσια, είναι πολύ θεσκευόμενοι άνθρωποι, παρόλα αυτά ή μάλλον ε, χάρη σε αυτό είναι άνθρωποι που ειρηνικοί. Ε, μιλούμε και για τις οικονομικές δυνατότητε τη χώρα. Δεν υπάρχουν οικονομικέ δυνατότητε. Η χώρα αυτή δεν έχει φυσικού πόρου πολύ συχνά πλημμυρίζει, ε, συμβαίνουν σεισμοί ε, και είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε δύο δύσκολους, δύστροπους γείτονες. Αν δεν υποστηρίξουμε οικονομικά και πολιτικά τον Νεπάλ, πιθανώς θα καταλήξει στη μοίρα του Θιβέτ. Κάτι που θα ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια για όλους μας. Ευχαριστώ. Θα κλείσει συζήτηση με τον Επιτροπή κύριο Νταλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Το αδιέξοδο στην πολιτική του Νεπάλ μας ανησυχεί και η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Στις 28 Μαΐου ήταν η προθεσμία ανακοίνωση του νέου συντάγματος. Βεβαίως απεφεύθη η κρίση με το να παραταθεί η προθεσμία για άλλο ένα έτος. Όμως πολλά επίμαχα ζητήματα εμποδίζουν τη διαδικασία. Όπως η φύση της ομοσπονδιακής δομής, η ενσωμάτωση των μαοικών ανταρτών και η ενοποίηση των δύο στρατών. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν η χώρα να πέσει σε ένα φαύλο κύκλο έλλειψης τάξεως και ασφάλειας. Δύο ζητήματα λοιπόν. Το Σύνταγμα και η ενσωμάτωση του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού περιπλέκουν την κατάσταση. Εάν δεν υπάρξει πραγματική διάθεση δούνε και λαβίνουν, ούτε και αυτό το ένα έτος θα αρκέσει. Η κατάσταση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, όπως ξέρετε επιτηρείται από αντιπροσωπεία της Αρμοσίας του ΙΕ στο Νεπάλ που έχει ε, ε, την αποστολή της για άλλο ένα έτος και η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχετική επίσης παρατηρεί την κατάσταση με τον πρόσφατο θάνατο Υπουργού και Προέδρου της ε, συνέλευσης ε, του Νεπάλ, του κυρίου Νεπάλ, ε, χάθηκε μία μορφή η οποία θα μπορούσε να επιλύσει διαφορές μεταξύ των κομμάτων και να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τον Νεπάλ να ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία. Οι δηλώσεις αρχηγών επικεφαλής αντιπροσωπιών και του ύπατου προσώπου καλούν όλα τα κόμματα να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Νεπάλ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Θα πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία θα οδηγήσει σε ειρήνη. Συλλογικά η Ένωση και τα κράτη-μέλη της ε, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της αναπτυξιακής βοήθειας του Νεπάλ η Κομισιόν συνεισφέρει στην ειρηνευτική διαδικασία με το να στηρίζει το ειρηνευτικό ταμείο του Νεπάλ 6 εκατομμύρια ευρώ πέρσι και 22 εκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί για το 2011 μέχρι στιγμής. Αυτά έχουν δοθεί για την συντήρηση των μαοικών μερών του Νεπάλ και για τους μισθούς των ανταρτών. Και ελπίζουμε λοιπόν όλος ο κόσμος να υποφελθεί από την ειρήνη όπως περιμένει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε συνεργασία με τα κρατημέλη κομισιών θα συνεχίσει όλες τις προσπάθειες διπλωματικές, πολιτικές και αναπτυξιακές για να συνεισφέρουν σε ένα δημοκρατικό και νεπάλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουν κατατεθεί συνολικά έξι ψηφίσματα από σοσιαλδημοκράτες, ε, πράσινους, ε, ελεύθερη ευρωπαϊκή συμμαχία, ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα αριστερών και φιλελεύθερων. Τελείωσε η συζήτηση και θα ακολουθήσει η ψηφοφόρια στο τέλος. Λοιπόν, θα συζητήσουμε κατόπιν το επόμενο θέμα της εκτελέσεις στη Λιβύη. Δίνω τον λόγο στον κύριο Τάνο και ένα λεπτό. Εγώ ποτέ δεν ήμουν απόλυτος ό,τι αφορά τη θανατική τιμή, αλλά μόνο θα πρέπει να ε, καταδικάζονται σε αυτή ε, στιγμή εγκληματίες όταν ε, έχουν υποστεί δίκαιη δίκη. Αλλά όμως δεν έχω εμπιστοσύνη στο λιβικό δικαστήριο.